Βλέπω κάτι πηγαδάκια στο κέντρο της αιθούσης. Colleagues, please, can we begin with our meeting? Συνάδελφοι, να ξεκινήσουμε με τη συνεδρίασή μας και όσοι δεν θέλουν να έχουν συμμετοχή μπορούν να απέλθουν. Έχουμε ακόμα καμιά δεκαριά ε, ανθρώπους που στέκονται εκεί σε αυτή τη ε, σειρά. Αποφασίστε αν θέλετε να λάβετε θέση ή να πάτε καμιά βόλτα έξω στο πάρκο που έχει περισσότερο χώρο. Ο Τόμας Τόμπε και εγώ θέλουμε να ξεκινήσουμε αυτή τη συνεδρίαση. Σας καλωσορίζω όλους. Να πω ευθύ εξ αρχή ότι θα περάσουμε στο σημείο 1 έγκριση τη ημερήσια διάταξη εφόσον δεν υπάρχουν σχόλια ή αντιρρήσει. Εγκρίνεται λοιπόν και πάμε στο σημείο 2 ανακοινώσεις του Προέδρου. Σε αντίθεση με άλλες συνεδριάσεις, σήμερα έχω μια σημαντική ανακοίνωση. Όλα τα μέλη της Επιτροπής Εξωτερικών Υποθέσεων, ιδιαίτερος όσοι ήταν και την περασμένη φορά μέλη, στην περασμένη θητεία, γνωρίζουν ότι ένα πολύτιμο τμήμα της Επιτροπής ΑΦΕΤ μας άφησε. Ένα πολύτιμο μέλος, η ε, Αμέλ Ντουό. Η Αμέλ Ντουό που καθόταν δίπλα μου επί χρόνια ήταν ε, υπεύθυνη για την ε, ΑΦΕΤ από τον Δεκέμβριο του 2015 μέχρι τον Σεπτέμβριο του 2019. Τέσσερα χρόνια βρέθηκε δίπλα μας. Επιβίωσε του Χέλμαρ Μπροκ ως πρόεδρου και μετά επιβίωσε και τον Μακάλιστερ ως πρόεδρο. Ακόμα πιο δύσκολο. Πρέπει να πω ότι με τα θλίψεις ακούσαμε τις ευχάριστες ειδήσει ότι θα φύγει, αλλά είχε μια πολύ ενδιαφέρουσα πρόταση. Τώρα είναι υποδιευθύντρια του Προέδρου του Κοινοβουλίου σας όλοι. Έχω καλέσει την ΑΜΕΛ σήμερα, εφόσον θέλει να πάρει μέρος στη συνεδρίαση της ΑΦΕΤ. Αμέλ, θέλεις να έρθεις ε, μπροστά και να σε ευχαριστήσουμε επισήμως για την πολύ καλή δουλειά που έκανες στην Επιτροπή ΑΦΕΤ την πρεμεσμένη τετραετία. So, merci Amel and good luck to you. And now we come to item number... Καλή τύχη λοιπόν Αμέλ. Πάμε στο σημείο 3. Μαζί με την Επιτροπή Ανάπτυξης και βάσει του άρθρου 58 στο σημείο 3 για τη δημιουργία ε, του εργαλείου συνεργασίας για τη γειτονία και την ανάπτυξη. Μια πολύ ενδιαφέρουσα νομοθετική πρόταση στα πλαίσια του πολυετούς νομοθετικού πλαισίου μέχρι το η ευρωπαϊκή βοήθεια προς τις τρίτες χώρες και τα ποσά που θα δαπανηθούν. Εδώ έχουμε μια κοινή ψηφοφορία για την έναρξη διαπραγματεύσεων με την Επιτροπή και το Συμβούλιο. Την πρώτη, τη θέση μας την εγκρινάμε σε πρώτη ανάγνωση από το Μάρτιο και θα είναι η βάση για τις διαπραγματεύσεις μας. Για τη διαδικασία μας τώρα υπάρχει ονομαστική ψηφοφορία ώστε να υπάρξει διαφάνεια στην όλη διενέργεια της ψηφοφορίας ε, ήταν προαιρετική αυτή η επιλογή βάσει του κανονισμού, αλλά θα ψηφίσουμε κατά αυτόν τον τρόπο και πρέπει να υπάρξει και πλειοψηφία όλων των μελών της Επιτροπής. 49 από 97 βουλευτές, διότι είμαστε 71 στην ΑΦΕΤ και 26 στην ΔΕΒΕ. Και μετά από την ψήφιση αυτή τη εντολή. Θα ψηφίσουμε και την, ε, διαπραγμάτευση, την έναξη διαπραγματεύσεων για το ε, εργαλείο αναπτυξική βοήθεια. Αυτά από την πλευρά μου και τώρα λόγο στον κύριο Τομπέ. Ευχαριστώ πολύ. Πολύ σύντομα μια και θέλουμε να εξοικονομήσουμε χρόνο, να σας πω πως από την πλευρά της ΔΕΒΕ επιβεβαιώνω πως ε, είναι ένας ε, φάκελος κομβικός και για τις δύο επιτροπές και θα καθορίσει την οικονομική στήριξη που θα προσφέρουμε εκτός συνόρων τα επόμενα χρόνια. Περιμένουμε λοιπόν με χαρά τις διαπραγματεύσεις που θα ξεκινήσουν το συντομότερο δυνατόν και ελπίζουμε πως ήδη μέσα στο μήνα, έτσι ώστε η διαφάνεια και η συμμετοχή όλων των επιτροπών ε, και οι ενημερωτικές συναντήσεις από τους συνεισηγητές θα γίνουν και θα οργανωθούν στα πλαίσια αυτής της κοινή ε, και δημόσιας προσπάθειας που θα κάνουμε. Πολύ ωραία. Ευχαριστώ πολύ, Τόμας. Μπορούμε λοιπόν να συνεχίσουμε με την ψηφοφορία. Τι ωραία. Για τις, τις σημειώσεις του Προέδρου που διαβάζω, λέει πως δεν θα γίνει άλλη συζήτηση λόγω ε, έλλειψης χρόνου. Οπότε μην τολμήσει κανείς να ζητήσει το λόγο. Περνάμε λοιπόν στην πρώτη ψηφοφορία. Είναι ηλεκτρονική. Άρχεται. Ένα συνάδελφος δεν έχει ψηφίσει. 87 out of 87. The vote is closed. Ωραία λοιπόν, πέρα τη ψηφοφορία, 87 στου 87 ψήφισαν, εγκρίνεται 72-15. We have a problem. Υπάρχει πρόβλημα. Okay, could a technician take care of that? Παρακαλώ να πάει ένας τεχνικός να το διορθώσει. Εγκρίθηκε 72-15. Μπορούμε να περάσουμε στο σημείο 4. Πρέπει να αλλάξουμε το σύστημα τώρα γιατί ψηφίζει μόνο η ΑΦΕΤ. So, item number για το 4 λοιπόν, μόνο τα μέλη της ΑΦΕΤ, όσοι ανήκουν στην ΤΕΒΕ δεν ψηφίζουν, βγάλτε τις κάρτες σας. Great. So, colleagues, item number four. Στο 4 λοιπόν, η απόφαση για διοργανικές διαπραγματεύσεις ε, στο ΙΠΑ, το εργαλείο αυτό για την προενταξιακή στήριξη. Μόνο τα μέλη της ΑΦΕΤ θα ψηφίσουν. Ζόφκο και τον Νίνο Πίτσουλα είναι οι δύο συνεισηγητές, ΕΛΚ και Σοσιαλιστές και για να εγκριθεί η απόφαση αυτή χρειάζεται μια πλειοψηφία των 71 μελών της ΑΦΕΤ, δηλαδή τουλάχιστον 36 υπέρ άρθρο 72 θα αποτελέσει την εντολή αυτή η πρώτη ανάγνωση για τις διαπραγματεύσεις. Άρα λοιπόν ψηφίζουμε, άρχεται η ψηφοφορία. Περισσεύει ένας πράσινος. Now there's one too much on. Τώρα περισσεύει και ένας από τη Ρινιού. This looks like an EPP point of view. Νομίζω ότι αυτή είναι η άποψη του ΕΛΚ ότι περισσεύουμε. Όχι, δεν περισσεύεται επειδή το πιστεύουμε, περισσεύεται επειδή το λέει ο υπολογιστή. Λοιπόν, ένας από τους πράσινους και ένας από τους Ρινιού, παρακαλώ να βγάλετε την κάρτα σας. Εντάξει, τώρα είμαστε όσοι πρέπει. 67 out of 73. 67 από τους 73 έχουν ψηφίσει. Έξι συνάδελφοι της ΑΦΕΤ ξεχαστήκατε. Θέλετε, μπορείτε, προλαβαίνετε. Okay, now I need one more going down. Problem is that. Would you share your technical information? It's 71... μέλη έχει η ΑΦΕΤ και το μηχάνημα μετράει 72 κάρτες. Ένας περισσεύει, αλλά δεν μας λέει ποιος περισσεύει. Ποιος παριστάνει ότι είναι μέλος της ΑΦΕΤ εδώ. Και τώρα μείνανε 6 οι πράσινοι, αλλά πρέπει να είμαστε 7. Άρα πάλι κάπου κάνει λάθος το μηχάνημα. Τώρα πέσαμε στους 70. Αλλά μόνο οι 66 έχουν ψηφίσει. Now we're 71 and now... No, now there's one green too much. Eh? Πάλι περισσεύει ένας πράσινος. okay, no. We close the vote. So we, we close the vote. Πέρας της ψηφοφορίας. And the result is 59 to 8, so... 59-8 το σκορ, άρα εγκρίνεται. Then we come to item number 5. Περνάμε στο 5 κοινή ψηφοφορία με την ΤΕΒΕ και σε συνεργασία με την Υποεπιτροπή για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα. Θα ψηφίσουμε λοιπόν για τον περιορισμένο κατάλογο των υποψηφίων για το βραβείο Ζαχάροφ. Αυτό θα γίνει και κλεισμένον των θυρών, οπότε μόνο τα εγκεκριμένα μέλη ή αξιωματούχοι του Κοινοβουλίου και οι ε, υπάλληλοι θα είναι παρόντες. Οι υπόλοιποι παρακαλώ να εγκαταλείψετε την αίθουσα. Και όσοι είστε εδώ παρακαλώ